So, once Mr. Rosati here, we start with point. Ήρθε λοιπόν ο κύριος Ροζάτη, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε την ε, παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών εφαρμογή των προτεραιοτήτων του υλοποίηση των προτεραιοτήτων για το 2015. Έχετε το λόγο κύριε Ροζάτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ζητώ συγγνώμη, περίμενα να είμαι στην ώρα μου γιατί προβλεπόταν η έναρξη τη συζήτηση του θέματος 9 και 4. Ο πρόεδρο έχετε δίκιο. Απλά λίγα δευτερόλεπτα μου χρειάστηκαν για να διεκπαιρώσω τα πρόταση με τις μερισιάς διάταξη. Κύριο Ροζάτη, η έκθεση λοιπόν αφορά το φετινό Ευρωπαϊκό Εξάμεινο 2015 και βασίζεται σε διάφορα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου. Το πρώτο και σημαντικότερο ίσως είναι η σύσταση της Επιτροπής για Σύσταση του Συμβουλίου σε σχέση με τη συστάσεις αναχώρα για το 2015. Αλλά φυσικά βασιζόμαστε σε μεγάλο βαθμό και στα προηγούμενα έγγραφα. Έχω και εγώ συντάξει νωρίτερα φέτος μια έκθεση για την επισκόπηση για την ανάπτυξη το 2015 και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρήση ευελιξίας ό,τι αφορά την ερμηνεία του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Η έκθεση υποδιέρεται σε τέσσερα τμήματα. Στο πρώτο τμήμα εκφράσουμε τη σύμφωνη γνώμη με τις απόψεις της Κομισιόν ε, για την εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης της Ένωσης, ιδίως στην υπέρχη της Ευρωζώνης. Βλέπουμε με ικανοποίηση ότι με βραδείς ρυθμούς ε, η ανάκαμψη επανέρχεται, αν και τα θεμελιά της είναι ακόμη αρκετά ευάλωτα. Με βάση όμως τις αρινές ε, εκτιμήσεις, η ανάπτυξη θα επιταχυνθεί για, ε, το χρόνο 2,1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2,1% στην Ευρωζώνη και αυτό είναι μια θετική εξέλιξη, διότι σηματοδοτεί κατά πάσα πιθανότητα την επιστροφή της Ευρωζώνης για πρώτη φορά από το 2009 στον δρόμο της Συμφώνου Σταθέρτας και Ανάπτυξης. Επίσης, στηρίζουμε και συμμεριζόμαστε τη νέα προσέγγιση την οποία ανέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν διατύπωσε τις φετινές συστάσεις αναχώρα. Αυτή η νέα προσέγγιση συνίσταται, κατά κύριο λόγο, στην εστίαση σε πολύ σημαντικές προτεραιότητες και προκλήσεις στο πλαίσιο αυτών των συστάσεων αναχώρα. Και αυτό είναι μια καλοδεχούμενη αλλαγή, διότι δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να εστιάσουν πραγματικά στις σημαντικότερες προτεραιότητες. Ταυτόχρονα, σημειώνουμε με ανησυχία ότι ο βαθμός δέσμευσης που επιδεικνύουν τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των συστάσεων αναχώρα είναι ανεπαρκής. Δηλαδή, υπάρχουν χώρες περισσότερο δεσμευμένε στην εφαρμογή των συστάσεων αναχώρα, πολλά άλλα κράτη-μέλη όμως εξακολουθούν να υπολείπονται. Κατά μία έννοια, θεωρούμε ότι αυτό συνιστά την επάρκεια του όλου συστήματος τη οικονομική διακυβέρνησης. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα χρειαστεί να επεξεργαστούμε συγκεκριμένα μέτρα για να καταστούν πιο δεσμευτικέ οι ανά χώρα. Το δεύτερο τμήμα αφορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη. Ευθυγραμμιζόμαστε και εδώ σε πολύ μεγάλο βαθμό με την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σημειώνουμε με ανησυχία ότι η ανεργία παραμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα ε, στα κράτη-μέλη. Βέβαια η κατάσταση είναι διαφορετική από τη μια χώρα στην άλλη. Βλέπουμε κάποιες διαφορές. Επίσης χαιρετίζουμε την ε, έναρξη ισχύω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Σημειώνουμε επίσης με ικανοποίηση ότι έχουμε λιγότερα κράτη-μέλη στη διαδικασία δημοσιονομικού ελλείμματος. Παρ' όλα αυτά, όσες χώρες παραμένουν στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας ε, πρέπει να αναβαθμίσουν τις προσπάθειές τους για να εξηγιάνουν ε, τα δημοσιονομικά τους. Οι συστάσεις αναχώρα δείχνουν ότι υπάρχουν ακόμη οικονομικές ανισορροπίες ε, σε διάφορες χώρες, οι οποίες επιμένουν. Και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να βελτιώσουν τις εθνικές τους πολιτικές για να διορθώσουν τις ανισορροπίες αυτές. Όπως είπα, στηρίζουμε τη νέα προσέγγιση της Κομισιόν που δεν συνίσταται μόνο στην εστίαση σε βασικές προτεραιότητες ολιγάριθμες, αλλά συνίσταται και στην επιτάχυνση του χρονοδιαγράμματος. Αυτό το βλέπουμε με την παρουσίαση των συστάσεων αναχώρα, οι οποίες συστάσεις υποβάλλονται τρεις μήνες νωρίτερα. Και αυτό είναι θετικό. Δίνει στις χώρες πιο πολλά χρονικά περιθώρια για να αφομοιώσουν τις συστάσεις, ε, για να έχουν διαβουλεύσεις με τους διαφόρους ε, φορείς και έτσι να προετοιμαστούν καλύτερα για την υλοποίηση αυτών των συστάσεων. Οι συστάσεις αναχώρα χώρα το 2015 είναι οργανωμένες γύρω από τέσσερις βασικές προτεραιότητες. Η πρώτη προτεραιότητα είναι η ανάγκη επιτάχυνσης των επενδύσεων. Εδώ στο πλαίσιο και αυτών των συστάσεων αλλά και στο πλαίσιο άλλων εγγράφων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαβάζουμε ορισμένες συστάσεις. Συγκεκριμένα, βελτίωση της πρόσβασης ε, ιδίως των ΜΜΕ ε, στη χρηματοδότηση για τόνωση των επενδύσεων ανά την Ευρώπη. Δεύτερη βασική προτεραιότητα. Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος που είναι βασικός παράγοντας για τη βελτίωση των επενδύσεων στην Ένωση. Στην έκθεσή μας λοιπόν τονίζουμε και εμείς ε, τη σημασία να έχουμε και τους ε, κατάλληλους ε, κανονισμούς. Τρίτη προτεραιότητα, κάτι που επανέρχεται έμφαση στην ανάγκη συνέχισης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ιδίω αγορές προϊόντων και υπηρεσιών. Στόχος είναι η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταστεί πιο ανταγωνιστική. Επιπλέον, ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στον τομέα αυτό είναι φυσικά η έμφαση για την καθιέρωση της ενέας ψηφιακής αγοράς. Τέταρτη προτεραιότητα, πολιτικές απασχόλησης. Πολιτικές απασχόλησης οι οποίε αφενός θα οδηγήσουν σε καλύτερε πιο ποιοτικέ θέσει εργασία. περισσότερες θέσεις εργασίας που θα προσφέρουν και υψηλότερε απολαβές όμως ταυτόχρονα και η κοινωνική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βελτιωθεί. Στο τελευταίο τέλος τμήμα της έκθεσης διατυπώνουμε ορισμένες συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως προανέφερα, ζητούμε από τα κράτη-μέλη τα οποία ε, είναι στο πλαίσιο των διαδικασιών μακροοικονομικών ισορροπιών να ε, κάνουν περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να συμμορφώνονται με τους κανόνες ότι αφορά τα δημόσια οικονομικά τους. Επίσης τονίζουμε το ρόλο των ευέλικτων αγορών εργασίας για την καταπολέμηση της ανεργίας και ιδίως της ε, ανεργίας των νέων και των μακροχρόνια ανέργων. Μια άλλη σύστασή μας είναι να βελτιωθεί η ιδιοκτησία, η ιδιοποίηση θα έλεγα. Γιατί τα κράτη-μέλη δεν εφαρμόζουν τις συστάσεις αναχώρα με την ίδια ένταση, αν μπορώ να το πω έτσι. Δεν τις έχουν ενστερνιστεί όλες στον ίδιο βαθμό. Επίσης, παραλαμβάνουμε την έκκλησή μας προς την Κομισιόν να εξορθολογήσει περαιτέρω τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμείου. Υπήρξαν βελτιώσεις σίγουρα φέτος, παρόλα αυτά, ίσως να είναι ακόμη υπερβολικός αριθμός των εγγράφων, τα οποία κυκλοφορούν στο πρώτο ήμιση της χρονιάς, επιβάλλοντας ακόμη μεγαλύτερο φόρτο εργασίας. Σύγκληση, εκθέσεις σύγκλησης, σταθεροποίησης, εθνικά προγράμματα, μέσα σε τρεις-τέσσερις μήνες. Είναι δύσκολο να μην υπάρξουν ε, ασυνέπειες μεταξύ των εγγράφων. Άρα θα πρέπει να υπάρξει περαιτέρω εξορθολογισμός αυτής της διαδικασίας. Ζητούμε επίσης τα καταστροφικά ε, επίπεδα χρέους να μειωθούν γιατί συνιστούν σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξη τόσο στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα βέβαια. Επίσης, υποστηρίζουμε και ορισμένες συστάσεις των πέντε προέδρων στην εκθεσή τους. Το έγγραφο αυτό νομίζουμε ότι είναι ένα σημαντικό έγγραφο γιατί ανοίγει τη συζήτηση για διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη. Λίγο πολύ αυτά είχα να πω. Προσβλέπω βέβαια στα σχόλια και στις παρατηρήσεις των συναδέλφων, κυρίως από τους σκιώδεις συζητητές των άλλων πολιτικών ομάδων και αναμένω ότι θα έχουμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση κατά την περαιτέρω εκπόνηση του σχεδίου έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Ρωσάτη, θα ήθελα τώρα να δώσουμε το λόγο στους σκιώδεις συγητές ξεκινώντας από τους σοσιαλδημοκράτες. Παρακαλώ. Ε, θα ήθελα να ξεκινήσω συγχαίροντας τον κύριο Ρωσάτη για μια πολύ καλή και στοχευμένη έκθεση η οποία έχει επίσης και το πλεονέκτημα ότι καταδεικνύει την ουσία. Βεβαίως ενδέχεται αυτή την έκθεση θα έλεγα να παραλείπονται κάποια θέματα τα οποία για μας είναι πολύ σημαντικά. Όσον αφορά τις συστάσεις αναχώρα θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για να επιτευχθεί ο στόχος της ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να καταγραφεί η απόδοση, η οικονομική απόδοση σε κάθε χώρα και αυτές οι συστάσεις αναχώρα πρέπει επίσης να αξιολογηθούν με κριτικό πνεύμα. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται, επειδή δεν υπάρχουν ε, άλλες ε, δομές, ε, θα πρέπει να αναπτυχθούν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως, αυτά που προτείνονται, πρέπει να πω, δεν είναι και απαραίτητα αδιαμφισβήτητα. Έχουν γίνει και κάποια λάθη. Παραδείγματο χάρη, φαίνεται ότι υπάρχει μια πλουστευμένη άποψη ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις έχουν μηχανική και αυτόματη ανάπτυξη στις θέσεις απασχόλησης και στην ανάπτυξη. Ε, βέβαια, αυτό σημαίνει ότι αν γίνουν αλλαγές στην αγορά εργασίας όταν υπάρξουν θέσει απασχόληση δεν σημαίνει ότι θα μετακυληθούν αυτόματα από τη μία χώρα στην άλλη. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν εναλλακτικέ λύσει και είναι πιο αποτελεσματικό να σταθεροποιούνται οι οικονομίες και να ε, προκαλείται εκεί η ανάπτυξη. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των παλαιότερων συστάσεων αναχώρα, αυτέ πρέπει να αξιολογηθούν και ίσω ε, θα πρέπει να εξετάσουμε και τι κοινωνικέ επιπτώσει των συστάσεων αναχώρα που εγκρίθηκαν κατά το παρελθόν. Για πέρυσι ας πούμε άκουσα ε, κριτική για το ότι δεν υπήρχε κάποια κοινωνική ευαισθησία μεταξύ άλλων σχετικά με αυτές τις συστάσεις και πιστεύω ότι αυτή η κριτική είναι δικαιολογημένη. Εξίσου σημαντικό είναι και αυτό που λέγεται ότι πολλές συστάσεις αναχώρα χρησιμοποιούν άκαμπτα κριτήρια, λαμβάνουν υπόψη τους τις τοπικές συνθήκες και αυτό οδηγεί σε ένα άλλο πολύ κρίσιμο θέμα ότι παρότι η γενικότερη στόχη είναι επιτευχθεί ε, σύγκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατ' ουσίαν η απόκληση μεγαλώνει και δεν υπάρχει ακόμα ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο να μπορούν να ενταχθούν αυτές οι τοπικές και άλλες διαφορές και εξάλλου η Οικονομική και Νομισματική Ένωση πολύ ισχυρή μετατραπεί σε μία ένωση μεταφοράς πόρων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι μία ένωση όπου μεταφορά οικονομίες εποφελούνται από άλλες που είναι πιο ισχυρές. Και αυτό προκαλεί μία συστηματική μεταφορά πόρων από κάποιες περιοχές σε άλλες περιοχές και αυτό γίνεται μέσα από το εμπόριο και τις οικονομικές ροές. Οι συστάσεις χώρα. δεν μπορεί να είναι το σωστό εργαλείο για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Η κατάσταση στην Ελλάδα δείχνει ότι εγκυμονούν και άλλοι περαιτέρω κίνδυνοι αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν υπάρξει μείωση της οικονομικής απόκλησης, η αποτελεσματικότητα των συστάσεων χώρων θα συνεχίσει να είναι προβληματική. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε, Χορ, κύριε Πρόεδρε. Εκ μέρους της ECR παρακαλώ, του κόμματο των Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ισηγητά, νομίζω ότι το σχέδιο ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση και επίσης ε, θεωρώ ότι μπορούμε να στηρίξουμε τις προτάσεις σας. Αλλά επιτρέψτε μου να κάνω και κάποιες ε, παρατηρήσεις. Φυσικά και πρόκειται για τη συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, πρόκειται για την έκθεσή μας. Σημείο υπαριθμών 4. Στο σχέδιο πρέπει να σας πω δεν συμφωνώ με τον εισηγητή. Δεν συμφωνώ όσον αφορά την εφαρμογή των ε, συστάσεων αναχώρα και αυτά στο πλαίσιο ενός ε, δίκαιου πλαισίου. Δεν είμαι πεπισμένος ε, ότι θα πρέπει να είναι αυτή η διατύπωση. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν κίνητρα για τις ε, χώρες έτσι ώστε να εφαρμόζουν τις μεταρρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο. Πάμε τώρα στο σημείο υπαριθμών 5. Πιστεύω ότι ακριβώς όταν πρόκειται για τη ζώνη του ευρώ, οι χώρες σε αυτή τη ζώνη αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα. Θεωρώ όμως ε, ότι το που εξάλλου ε, θα πρέπει να υπάρξει μια αναδιατύπωση για να είναι σαφέστερο το σημείο αυτό. Πάμε τώρα στο σημείο υπαριθμών 15 στην έκθεση. Συμφωνώ όσον αφορά τις αγοράς εργασίας, για την αντιμετώπιση της ανεργίας, όμως οφείλουμε να επισημανούμε ότι και ξέρετε μερικές φορές εδώ γίνεται εκμετάλλευση του θέματος, ε, γίνεται εκμετάλλευση, προκύπτει εκμετάλλευση εκ μέρου των εργοδοτών και δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Ως εκ τούτου οφείλουμε να μεριμνήσουμε έτσι ώστε να μην υπάρξει ε, εκμετάλλευση και κακοδιαχείριση και από τις ε, δύο πλευρές. Και επιτρέψτε μου και μία παρατήρηση για το σημείο υπερθμών 7. Ε, θέλω να σας πω όσον αφορά το σημείο υπερθμών 7, όπου γίνεται λόγος ε, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Απεντήσεων, πράγματι έχει δίκιο, αλλά πρέπει να είστε και λίγο προσεκτικοί όσον αφορά τους στόχους αυτού του Ταμείου στην ε, έκθεση πρέπει να γίνεται λόγος και για συντονισμό των ε, μεταρρυθμίσεων αλλά εν πάση περιπτώσει σας είπα και αυτής εξ αρχής ότι αυτές ήταν ε, κάποιες ε, μικρές παρατήσεις που είχα να κάνω τώρα δεν έχω να κάνω σημαντικότερες παρατήσεις. μου αρέσει πολύ η έκθεση και συγχαίρω τον εισηγητή για την πάρα πολύ καλή δουλειά του σας ευχαριστώ πολύ Ευχαριστώ πάρα πολύ Ταβάρ έχει το λόγο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω μετά τις διακοπές. Εδώ είμαστε λοιπόν, συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και κάπου το έχουμε ξαναδεί το έργο. Πριν εξηγήσω τι εννοώ, να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον εισηγητή για το σχέδιο έκθεσης. Νομίζω πως αντιμετωπίζει το ζήτημα με τον σωστό τόνο και φύγει τα σωστά ζητήματα. Λοιπόν, θα σκεφτώ κάποιες ε, βελτιώσεις και θα καταθέσω κάποιες ανάλογες ε, τροπολογίες. Δεν έχω πιστεί ιδιαίτερα για το θέμα του καλύτερου συντονισμού της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με το, με το EDP, καθώς ε, το πρώτο κομμάτι είναι στο πλαίσιο του προληπτικού σκέλους. Επίσης, η ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου πρέπει να πάει χέρι-χέρι με μια μεγαλύτερη έμφαση στην διαφάνεια ιδιαίτερα όσον αφορά την ε, μεθοδολογία η οποία εφαρμόζεται καθώς αυτό δύσκολα γίνεται αντιληπτό άρα θα πρέπει να γίνουν τα πράγματα πιο ξεκαθαρά και μετά να δημοσιευτούν στο σύνολό τους. Επίσης θα θέλαμε να δούμε την οικονομική ανάλυση της ε, Κομισιόν για να ξέρουμε δημοσίως ε, το τι γίνεται. Ε, τώρα για την παράγραφο 13, τι εννοεί ο εισηγητής, ότι ο αυτόματος θα πρέπει να κάνει το έργο ή ζητάμε εδώ πέρα μια ενεργή ε, δημοσιονομική πολιτική. Μοιάζει σαν ε, να βγήκε από την γενική θεωρία που δημοσιεύτηκε το 1936 και όχι να ταιριάζει το 2015. Τέλος, ε, τι, είπα, τι εννοούσα όταν είπα πως ε, είχαμε ξαναδεί το έργο. Υπενθυμίζω πως ε, τα κράτη-μέλη εφάρμοσαν μόνο 10% των συστάσεων αναχώρα και ίσως νομίζετε ότι δεν γίνονται χειρότερα τα πράγματα αλλά τελικά έπεσαν στο 7%. Ναι. Ε, βεβαίως, ναι, ναι, ε, ίσως η Κομισιόν να μας πει πως ε, τα νούμερα αυτά είναι λάθος. Αν όχι, θα ήθελα να μας εξηγήσει η Κομισιόν γιατί είναι τόσο χαμηλός ο αριθμός εφαρμογής των συστάσεων ε, αναχώρα και τι σκοπεύουν να κάνουν γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αναμένω τη συνεργασία με τον εισηγητή γιατί συνήθως είναι λογικός άνθρωπος και νομίζω πως θα επιτύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα στο τέλος. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μαρίζα Ματέης έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που άργησα. Δεν παρακολούθησα την αρχική παρουσίαση. αλλά για την έκθεση αυτή παρά το ότι έχω διαφορετική άποψη συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε ο εισηγητής κάπου το έχουμε ξαναδεί το έργο η έκθεση αυτή επιμένει στις ίδιες αποτυχημένες συνταγές και μάλιστα πάει και ένα βήμα παραπέρα και προφανώς δεν πρόκειται να λύσει κανένα από τα ουσιαστικά προβλήματα του ευρωπαϊκού εξαμήνου. Μιλάει για περαιτέρω επαγρύπνηση όσον αφορά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την εφαρμογή τους. Επιμένει στο να δοθεί ένα μέτρο αυτονομίας ε, στα Εθνικά Κοινοβούλια, αλλά δεν φτάνει σε αυτό το οποίο θέμενος κοινοβουλευτική δημοκρατία. Και ένα άλλο στοιχείο αυτής της έκθεσης, σε σύγκριση με τις ε, προηγούμενες είναι πως ανοίγει εδώ πέρα ένα παράθυρο για αύξηση επιτοκίων, κάτι το οποίο δεν ε, καταλαβαίνω. Εδώ πέρα ανοίγουμε ε, επικίνδυνες πόρτες δεδομένων των όσων έχουμε δει. Τώρα δεν θα τα πω όλα παράγραφο παράγραφο, αλλά θεωρώ πως υπάρχουν κάποια σοβαρά ερωτήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, Ε, υπάρχουν πράγματι κάποιες μακροοικονομικές ανισορροπίες και προκλήσεις, αλλά αυτά δεν θα αντιμετωπιστούν με γενικόλογες ε, αναφορές στο εξωτερικό χρέος, το οποίο διαφέρει από χώρα σε χώρα. Επίσης θα πρέπει να γίνει πιο λεπτομερής αναφορά στην υψηλή ανεργία και τις διαφορετικές κοινωνικές δυσκολίες ε, που υπάρχουν. Επίσης, ε, μιλάει για το χρέος χωρίς να γνωρίζει ότι η λιτότητα είναι μία από τις αιτίες της ε, μεγαλύτερης υπερχρέωσης ε, των χωρών. Παραδείγματος χάρη, μιλάει για αύξηση της πρόσβασης στις επενδύσεις, αλλά δεν αναφέρει το γεγονός ότι όπου έχει συμβεί κάτι τέτοιο, έχει συμβεί ακριβώς λόγω του ότι υποχώρησε η λιτότητα, όχι λόγω της ε, μεγαλύτερης ε, πρόσφορας ε, και ζήτησης επενδύσεων. Όπως είπα δεν θα αναφερθώ σε κάθε παράγραφο, αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμές το να αγνοούμε τις ελαφρές βελτιώσεις που έχουμε δει είναι λάθος. Επίσης όσον αφορά την αύξηση των δημοσίων επενδύσεων αυτό είχε θετικά αποτελέσματα και επίσης αγνοείται από την έκθεση. Τον επικεντρωνόμαστε μόνο στις αποτυχημένες πολιτικές του παρελθόντος είναι χονδροειδές λάθος και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να επαναλαμβάνουμε τα λάθη του παρελθόντος. Επιπλέον δεν υπάρχει καμία βελτίωση της ε, δημοκρατικής ε, λογοδοσίας, κάτι το οποίο οπωσδήποτε επιδεινώνει την ε, κατάσταση και ξυπακούεται πως ε, είμαστε πάρα πολύ επικριτικοί απέναντι σε αυτή την έκθεση. Εννοείται ότι θα καταθέσουμε τροπολογίες και η πολιτική γραμμή την οποία πρασιζόμαστε δεν είναι πολύ συμβατή με αυτή την έκθεση. Εν πάση περιπτώσει η έκθεση αυτή είναι πολύ σημαντική και ελπίζουμε πως είναι πάρα πολύ, και θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα για να το αφήσουμε να περάσει έτσι. Υπάρχουν ε, διαφορετικές ε, λύσεις που δεν αναφέρονται καθόλου από τον ε, εισηγητή. Αυτό το οποίο λοιπόν θέλουμε να κάνουμε πρώτα απ' όλα είναι να επιλύσουμε την κρίση μέσω της προώθησης της απασχόλησης, της προώθησης των εθνικών οικονομιών και της ενίσχυσης των δημοκρατικών επιλογών. Σας ευχαριστώ για τους πράσινους ορτασούν. Yes, bueno, Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το έργο του. Ελπίζω να έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Κάποια σχόλια για την έκθεση. Πρώτα απ' όλα, επειδή είναι η πρώτη έκθεση μετά τα συμβάντα του καλοκαιριού, όπου θα πλέον να ασχοληθούμε με την οικονομική ε, κατάσταση και εξελίξεις, δεν νομίζω ότι μπορούμε να παραλείψουμε τα προβλήματα με την επιβράδυνση της κινέζικης οικονομίας ε, και επίσης ε, ε, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Ξέρουμε ότι πολλές φορές, μάλλον μέχρι τώρα για να έχουμε ένα ισορροπημένο εξωτερικό ισοζύγιο, βασιστήκαμε σε κάποια μέτρα όπως ήταν η συγκράτηση των μισθών, και τα λοιπά. Και πρέπει να ίσως να τα αναθεωρήσουμε όλα αυτά. Στο, ο εισηγητής αναφέρεται στα προβλήματα ανεργίας που αντιμετωπίζει η Ευρωζώνη, μιλά για απαράδεκτα υψηλά επίπεδα, συμφωνώ να περιμένει ο εισηγητής ότι η ομάδα μας θα καταθέσει τροπολογίες ό,τι αφορά τι είδου εργασία έχει δημιουργηθεί με βάση τα μέτρα που προτείνονται από τις συστάσει αναχώρα, τι επιπτώσεις έχει αυτό σε ό,τι αφορά την εποχική εργασία και πόσο αποδυνάμωσε τις οικονομίες μας ε, ουσιαστικά αυτή ε, η προσέγγιση με αυτό το πολύ μεγάλο επίπεδο εποχικότητας και επισφάλειας της εργασίας και τα προβλήματα που δημιουργεί. Τέλος, ό,τι αφορά την απασχόληση, νομίζω ότι στο 15 σημείο ε, γίνεται μία αναφορά στα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή λόγω των υπερβολικά υψηλών επιπέδων κατώτατων μισθών. Νομίζω ότι είναι τελείως ε, λάθος η προσέγγιση αυτή και ελπίζω να μας στηρίξουν και άλλες ομάδες για να το ε, αλλάξουμε αυτό το σημείο όταν λέει υπερβολικά επίπεδα κατά το μισθό. Επίσης, μιλάτε για το ότι δεν είναι ισχυρά τα θεμέλια της ε, ανάπτυξης και συμφωνώ. Θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στις επενδύσεις. Καλύπτεται το θέμα, αλλά πρέπει να το τονίσουμε ακόμη περισσότερο. Και υπάρχει και η απαθή εσωτερική αγορά. Ε, είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. θα είναι πολύ λιγότερη η εξωτερική ζήτηση λόγω των διεθνών συνθήκων και γι' αυτό πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα. Σε ό,τι αφορά τώρα τις μεταρρυθμίσεις, χαίρομαι γιατί ο εισηγητή αναφέρεται ρητά ε, στους ε, στόχους ε, του ορίζοντα 2020 σε σύνδεση με τις τάσεις αναχώρα. Στις προηγούμενες εκθέσεις χρειάστηκε να πολεμήσει η ομάδα μου να συμπεριληφθεί αυτή η συσχέτιση. Χαίρομαι που ε, τώρα ε, το βλέπω στο κείμενο και όσοι ήθεστε ε, για τις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα επιμείνουμε στο scoreboard, στους δείκτες ενεργειακής απόδοσης, κοινωνικούς δείκτες, θα επιμείνουμε σε αυτή τη γραμμή γιατί έχει δεσμευτεί η Κομισιόν αυτό τον πίνακα, αυτό το scoreboard να τον κάνει πιο πλήρη η Κομισιόν και εμείς θα συνεχίσουμε να επιμένουμε. Συνεχίζω. Συμφωνώ, όπως είναι προφανές, με πολλά από τα σχόλια που έγιναν σε ό,τι αφορά το δημοκρατικό έλεγχο της όλης διαδικασίας. Και πιστεύω ότι εδώ υπάρχει ένα στοιχείο που δεν μπορούμε να παρακάμψουμε, ότι και οι κοινωνικοί ε, εταίροι ε, πρέπει να συμμετέχουν πολύ περισσότερο. Οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να παρεμβαίνουν, όπως γίνεται άλλωστε και με τον διαθροτικό διάλογο που γίνεται σε εθνικό επίπεδο. Γιατί να μην γίνεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί συστάσεις ανά χώρα. Γιατί όταν μιλάμε για έλλειψη οικειοποίησης και από τους κοινωνικού φορείς αλλά και από τα Εθνικά Κοινοβούλια, άλλο σημαντικό εταίρος, ε, αν αυτοί δεν συμμετέχουν, δεν μπορούμε να έχουμε πραγματικά σωστή διαδικασία Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Τρία ακόμη σημαίνει και ολοκληρώνω. Οι εσωτερικές ανισορροπίες ε, του ε, εξωτερικού ισοζυγίου το είδαμε και το καλοκαίρι με ε, χώρες με ρεκόρ πλεονάσματος ε, και αντίθετες ε, περιπτώσεις, αυτό, αυτή τη διαφορά πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Το χρέος που αναφέρει ο εισηγητής, ιδίως το 5, στην παράγραφο 5, έχουμε να αντιμετωπίσουμε τους επόμενους ε, μήνες τη διαδικασία, όπως όλοι περιμένουν τουλάχιστον, αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους. Υπάρχουν τα απαραίτητα εργαλεία και μέσα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είμαστε βέβαιοι γιατί είναι πολιτική γνωστή. Όλα αυτά πρέπει να αναφέρω και ολοκληρώνω με μία παράκληση στην ε, Επιτροπή για τα δικαιώματα της γυναίκας και ισότητα ε, φύλων. Έχουμε μία γνωμοδότηση κατά ε, παράδοση η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων δεν έχει επιδείξει και τόσο μεγάλη ευαισθησία για την ενσωμάτωση των τροπολογιών που αφορούν τη διάσταση του φύλου δεν τις έχει λάβει υπόψη τις, ε, αυτές τις τροπολογίες συνήθως ε, στα περιβαρπαϊκού εξαμήνου. Περιμένουμε τις τροπολογίες ε, της Επιτροπής Γυναικών και γιατί κανείς δεν έχει αξιολογήσει ή μελετήσει τον αντίκτυπο ε, τον ορισμένο τουλάχιστον από τις μεταρρυθμίσεις που προτείνονται για την ισότητα των φύλων. Παραδείγματο χάρη, μεταρρύθμιση τη αγορά εργασία. Έχουμε τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού. Στην Ισπανία, τη χώρα μου. Αυτά όλα επηρέασαν πολύ αρνητικά την κατάσταση τη ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Αυτά όλα πρέπει να τα αναλύσουμε. Αυτά θα συνεργαστούμε, ελπίζω, πολύ καλά με τον ε, εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ, Ερνέστ, λέει ο πρόεδρο. Ο κύριο Βάλιο από την ομάδα EFD. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ ευχαριστώ τον εισηγητή που μας παρουσίασε αυτό το κείμενο και επίσης ευχαριστώ και τους σκιώδης ε, γιατί είμαι σίγουρος ε, ότι θα συμβάλλουν και αυτοί στη συζήτηση. Όπως και στις ε, τελευταίες εκθέσεις, δυστυχώς η δική μου η ομάδα δεν συμφωνεί με την άποψη της πλειοψηφία και συμφωνούμε κατά τη με κάποιες από τις απόψεις που εκφράστηκαν από τους και ε, έχουμε λοιπόν τις δικές μας τις προτάσεις, τις οποίες και θα τις καταθέσουμε με τροπολογίες. Όσον αφορά τη στρατηγική της Κομισιόν, ότι για την ανάπτυξη πρέπει κανείς να βαθίσει σε διαρθρωτικές ε, αλλαγές και στη λιτότητα, όπως τα αναφέρει ο εισηγητής για να υπάρξει ανάπτυξη, εδώ δεν συμφωνούμε γιατί η πραγματικότητα έχει δείξει το αντίθετο. Δηλαδή αυτές οι προτάσεις απλά επιδίνωσαν την κρίση. Όσον αφορά τις ε, προτεραιότητες, των συστάσεων αναχώρα θα πρέπει να είναι ο γόνος κατά της απασχόλησης, αντιμετώπιση της στόχιας και αντιμετώπιση των ε, ε, οξυνόμενων διαφορών ε, και το αύξηση ή το άνοιγμα της ψαλίδας. Πρέπει λοιπόν να δοθεί σημασία στο να μην υπάρχουν μακροοικονομικές ανισορροπίες, κυρίως αυτές που προκύπτουν από υπερβολικά πλεονάσματα, γιατί αυτά οδήγησαν κατά κύριο λόγο στην οικονομική ανισορροπία και στην κρίση της Ευρωζώνης. Επίσης είναι απαραίτητο να καταγγείλουμε την αδράνεια της Κομισιόν, η οποία έχει αποφύγει να λάβει στοχευμένα συγκεκριμένες ε, προτάσεις και αλλαγές. Ε, θεωρώ ότι θα πρέπει κάπως ε, στην έκθεση αναφερθεί αυτό γιατί υπάρχουν σημαντικές ανισορροπίες οι οποίες απλώ οδηγούν στην επιδείνωση της κρίσης. Όσον αφορά τώρα στην ευελιξία την οποία ανέφερε και ο εισηγητής εμείς πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι τα περιθώρια της ευελιξίας που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία αυτά τα περιθώρια είναι ανεπαρκή. Δεν έχουν τα κράτη το απαραίτητο περιθώριο για να εφαρμόσουν αντικυκλικές πολιτικές. Ε, στην έκθεση επίσης αναφέρεται η θετική επίδραση της ευελιξίας των αγορών και δείχνουν όμως τα στοιχεία ότι οι αλλαγές που έχουν προαχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι μόνο αύξησαν την ε, ανεργία αλλά επιδίνωσαν γενικότερα την κατάσταση. Ε, η, κατά την άποψή μας η απελευθέρωση στην αγορά εργασίας ε, δεν οδήγησε σε ανάπτυξη. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα υποβάλουμε πάρα πολλές τροπολογίες. Τι να κάνω, λυπάμαι πάρα πολύ που είμαι τόσο επικριτικός, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η θέση μας. Ε, λυπάμαι πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ξεκινάει η διαδικασία Catch the Eye και θα ήθελα να ξεκινήσω από τον κύριο Μαριά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Uh, sorry. Μισό λεπτό λέει ο Πρόεδρος. Συγγνώμη κύριε Μαριά. Ε, δίνω το λόγο στη νέο σε ομάδα. Συνάδελφοι, σήμερα κάνουμε αυτή την συζήτηση για το όνειρο της ε, ενωμένης ε, υποτίθεται ευρωπαϊκής οικονομίας και όπως ε, λέει και το ρητό υπάρχουν μικρά ψέματα, υπάρχουν μεγάλα ψέματα και μετά υπάρχει και η στατιστική. Έτσι βλέπουμε ε, να μας μιλάνε εδώ πέρα για ανάπτυξη 2% του ΑΕΠ. να με συγχωρήσει ο αλλά Δυστυχώς ε, τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα όσο τα περιγράφει η Κομισιόν. Ε, γράφει δυσάρεστες αλήθειες στις συστάσεις ε, αναχώρα, ειδικά και για την χώρα μου και το Βέλγιο, δηλαδή από το οποίο κατάγομαι, υπάρχει μια μικρή όθηση στην ανάπτυξη, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις χαμηλές του πετρελαίου και βεβαίως η έλλειψη επενδύσεων οφείλεται στο βουνό του χρέους, του δημοσίου χρέους, το οποίο συνεχίζει να ψηλώνει και συνεχίζει άρα να καταστρέφει την εμπιστοσύνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο κοινό νόμισμα. Ο συντονισμός της ε, πολιτικής είναι επίσης ε, ένα μέσο το οποίο προσπαθεί να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα και να δώσει μία επίφαση αξιοπιστίας ε, για να μπορέσει να γεφυρώσει το κενό μεταξύ Νότιας και Βόρειας Ευρώπης όσον αφορά τα κοινωνικά. Κάτι το οποίο βεβαίω δεν θα καταφέρει και μετά αρχίζει να μας μιλάει για μια ομοσπονδιακή Ευρώπη και άλλα όνειρα θερινής ε, νυχτός. Δεν χρειάζεται κάτι ε, τέτοιο θα πρέπει απλά να αναπτυχθούμε σε ένα πιο σύνομο σπονδιακό πλαίσιο, ο καθένας με τις δικές του δυνάμεις και δυναμίες. Σας ευχαριστώ και με συγχωρείτε κύριε συνάδελφε Λοιπόν, τώρα περνάμε στο KTI. Ο κύριος Μαριάς και ο κύριος ε, Χέις έχουν ζητήσει τον λόγο. Κάποιος άλλος. Λοιπόν, κύριε Μαριά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση είναι πράγματι σημαντική. Να ε, ευχαριστήσω και τον εισηγητή για την παρουσίαση. Έχει θέσει ορισμένα θέματα, αλλά νομίζω ότι είναι ευκαιρία να συζητήσουμε επί της ουσίας. Πρώτα απ' όλα ε, τα σημεία 3 και 4 της εκθέσεως θέτουν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λειτουργήσει το περίφημο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι εδώ μιλούμε στη σφαίρα της οικονομικής πολιτικής. Επομένως από πλευράς αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μιλούμε για μια συντρέχουσα αρμοδιότητα και όχι αποκλειστική που σημαίνει ότι η κύρια ευθύνη για την άσκηση της οικονομικής πολιτικής ανήκει στα κράτη-μέλη και ο συντονισμός και η συζήτηση που κάνουμε εμείς και οι προτάσεις της Κομισιόν έχουν το στοιχείο της επιβοήθησης και όχι της επιβολής. Δυστυχώς έχει διαμορφωθεί ένα μοντέλο το οποίο είναι γραφειοκρατικό, επιβλητικό, προσπαθεί από τα πάνω να περάσει και να φέρει εντολές στα κράτη-μέλη και να μειώσει τις εξουσίες των εθνικών κοινοβουλίων. Ενώ πρέπει να συμβεί το αντίθετο. Οι εξουσίες ανήκουν στα κράτη-μέλη, στα εθνικά κοινοβούλια και εμείς εδώ ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πολύ περισσότερο η Κομισιόν συμβάλλουν σε μια συζήτηση προκειμένου να έχουμε ευμενή αποτελέσματα στην οικονομική ανάπτυξη των κρατών μελών. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέξουμε πώς διαρθρώνουμε το διάλογο που σημαίνει να δοθεί μεγαλύτερος ρόλος στα εθνικά κοινοβούλια που σημαίνει εδώ σε αυτό το φόρουμ να έχουμε μια συζήτηση και με μέλη των εθνικών κοινοβουλίων για να μπορέσει να προχωρήσει ε, μια ε, θετική παρέμβαση ε, επιβοήθηση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερο στοιχείο είναι να δούμε οι προτάσεις που κάναμε και αυτές που εφαρμόστηκαν τι αποτελέσματα είχαν. Διότι τελικά συζητούμε τι συστάσεις εφαρμόστηκαν αλλά δεν συζητούμε τα αποτελέσματα των συστάσεων. Τα οποία αποτελέσματα των συστάσεων δυστυχώς είναι δυσμενή για την οικονομική ανάπτυξη των κρατών μελών. Επιμένει η Κομισιόν και βλέπω και η πλειοψηφία εδώ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ένα μοντέλο αποτυχημένο. Επιμένει στη λιτότητα, επιμένει στο να μην αντιμετωπίζει το ζήτημα του δημοσίου χρέους, επιμένει σε πολιτικές αποδιάρθρωσης των αγορών εργασίας, επιμένει σε χαμηλούς μισθούς, ενώ το αντίθετο εμείς πρέπει να δώσουμε έμφαση σε επενδύσεις εντάσσεως τεχνολογιών, σε επενδύσεις οι οποίες θα αναπτύξουν πραγματικά την ευρωπαϊκή οικονομία σε μια άλλη κατεύθυνση. Δεν μπορεί να κινεζοποιηθεί η ευρωπαϊκή οικονομία αν θέλουμε να έχουμε αποτέλεσμα. Τρίτο θέμα, σημαντικό, ανεργία. Υπήρξαν τόσες παρεμβάσεις, τόσες συστάσεις. Ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα, το έχετε δει. Τεράστια ανεργία ιδίω των νέων στην Ελλάδα, την Ισπανία και σε άλλες χώρες για την Ελλάδα, πρέπει να σας πω ότι το μοντέλο έχει αποτύχει. Και αυτό το είδατε με αποτέλεσμα τις συζητήσεις που είχαμε το τελευταίο εξάμεινο με αφορμή την Ελλάδα. Όλοι οι δείκτες απέτυχαν. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε 240 δισεκατομμύρια ευρώ ως δάνεια, τελικά ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Ήταν να έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους και 40% του ελληνικού λαού να ζει στη φτώχεια δεν πρέπει να καταλάβει η ίδια η Κομισιόν, το Διεθνές Ομισματικό Ταμείο, η Τρόικα ότι έχει αποτύχει αυτή η πολιτική. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Άρα λοιπόν πρέπει να πάμε σε άλλη κατεύθυνση. Αλλά και το νέο μνημόνιο που επιβλήθηκε, στο οποίο συμφώνησε και ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ανεξάρτητοι Έλληνες και πλέον οι νέο μνημονιακές δυνάμεις θα φέρουν δυσμενή αποτελέσματα. Φορομπηκτική πολιτική, ε, δεν αντιμετωπίζουν το θέμα της ανεργίας. Άρα πρέπει να αλλάξει η κατεύθυνση και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε με δύο σύντομες παρατηρήσεις. Το θέμα του χρέους. Το αναφέρουν ε, πράγματι ο εισηγητής στα σημεία 5, 13 και 18. Αλλά δεν λέει την πρόταση. Η πρόταση για την ρύθμιση του χρέους πρέπει να είναι η διαγραφή του επονίδης του χρέους. Πρέπει να είναι το κούρεμα αυτό το οποίο είπε η κυρία Μέρκελ για την Ελλάδα είναι μια καραμέλα. Δηλαδή είπε ότι δεν θα γίνει κούρεμα, είπε ότι δεν θα μειωθούν τα επιτόκια και απλά θα γίνει επιμήκυνση. Μα δεν είναι αυτό η λύση, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και τις άλλες χώρες. Άρα λοιπόν αν αυτά δεν αντιμετωπιστούν και δεν συζητηθούν, νομίζω ότι δεν μπορούμε να έχουμε ευμενή αποτελέσματα για την οικονομική εξέλιξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Indeed, Mr. Σα ευχαριστώ. Τέλο τον λόγο έχει ο κύριο Χέι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε να συγχαρώ τον συνάδελφό μου για την εξαιρετική έκθεση. Νομίζω πως ε, έχει αναφέρει όλα τα σημαντικά στοιχεία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και νομίζω πως τα μέλη της Επιτροπής μας πρέπει να δουν την διαδικασία αυτή ως ένα σημαντικό όχημα μεταρρύθμιση στα κράτη-μέλη και να στηρίξουν την διαδικασία ως ευρωβουλευτής από μικρή χώρα, μία μικρή χώρα όμως η οποία πέρασε τρομερή οικονομική κρίση θα έλεγα το εξής ε, καταφέραμε να δούμε σημαντικά επίπεδα ανάπτυξης ε, και απασχόλησης ε, λόγω ακριβώς των οικονομικών μεταρρυθμίσεων που έγιναν και νομίζω πως ε, και για άλλες χώρες οι οποίες ε, ε, έχουν δει σοβαρές ανισορροπίες αυτό είναι κάτι το σημαντικό. Δεν θα δούμε βελτιώσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση αν δεν γίνουν μετα... μεταρρυθμίσεις διαρθρωτικές και ακριβώς οι συστάσεις αναχώρα είναι σημαντικό κομμάτι αυτής της διαδικασίας ε, γιατί ασκούν πίεση και ορθώς στους πολιτικούς εντός των κρατών μελών για να βρουν το σωστό μείγμα πολιτικής. Νομίζω πως ε, το κοινό, ειδικά στις χώρες που έχει περάσει, έχουν περάσει αυτό το τεράστιο να ζητούν μια πιο κριτική αξιολόγηση της εγχώριας πολιτικής, ε, ζητούν περισσότερο έλεγχο και εποπτεία και αν η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μπορεί να βοηθήσει τόσο το καλύτερο. Στην περίπτωση της Ιρλανδίας δεν συμμετέχουμε. Βγήκαμε από το οικονομικό πρόγραμμα το 2013 και καλωσορίζουμε το ότι οι συστάσεις δίνουν βάρος στα δημόσια οικονομικά, την υγεία, τα σταγαστικά δάνεια και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Θα πρέπει οι στάσεις αυτές ε, να είναι το μέτρο με το οποίο θα κρυφτεί οποιαδήποτε Ιρλανδική κυβέρνηση. Όπως είπα έχουμε δει ήδη σημαντικές βελτιώσεις οι οποίες είναι αποτελέσματα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έκανε η Ιρλανδική κυβέρνηση. καλοδεχούμενες και οι παρατηρήσεις που αφορούν τις φετινές αλλαγές. Είναι σημαντικό ότι θα δημοσιευτούν τρεις μήνες νωρίτερα οι συστάσεις αυτές. Και για αυτό το οποίο είπε μόλις ο κύριος Μαριάς, όταν τα εθνικά κοινοβούλια συζητούν τις εθνικές συστάσεις, θα πρέπει και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είμαστε μέσα σε αυτή τη συζήτηση. Τη στιγμή που γίνεται η συζήτηση, όχι εκ των υστέρων, όπως γίνεται τώρα. Οπότε ελπίζω αυτοί οι τρεις μήνες παραπάνω που έχουμε, μια που δημοσιεύονται νωρίτερα οι συστάσεις χώρα θα μας βοηθήσουν στη συζήτηση αυτή. Λοιπόν, κάποιες παρατηρήσεις για τις ε, επενδύσεις και συμφωνώ εδώ πέρα με τους συναδέλφους. Οι χώρες που έχουν περάσει πρόγραμμα όπως η δικιά μου που είδαν 20 έω 25% μείωση των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα υπάρχει ένα επιπλέον βάρος ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει αυτές τις χώρες ε, που πέρασαν πρόγραμμα Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ελλάδα και τις λοιπές που έχουν δει τόση μεγάλη μείωση των ιδιωτικών επενδύσεων. Πρέπει λοιπόν οι επενδύσεις να χρησιμοποιηθούν σε αυτές τις χώρες και μάλιστα με τρόπο εμπροστοβαρή. Κατόπιν, οι συστάσεις αναχώρα κοστίζουν λεφτά. Έχω πει πως πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον προπολογισμό της Ένωσης για να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη για να κάνουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Γιατί αν προσπαθεί κανείς να κάνει τα πράγματα διαφορετικά υπάρχει κάποιο κόστος αρχικό στην διαδικασία αυτή. Και ξέρω πως το έχει πει και ο κ. Σόιμπλε τελευταία, πως πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο προπολογισμό της Ένωσης για να ενθαρρύνει τις χώρες για να υιοθετήσουν αυτές τις συστάσεις αναχώρα. Κάτι άλλο. Ε, οι συνάδελφοι αναφέρθηκαν στην αβεβαιότητα του καλοκαιριού, τις δυσκολίες που υπάρχουν στην Κίνα και τα προβλήματα που θα δημιουργήσει αυτό ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπως το κινέζικο παράδειγμα σημαίνει ότι πρέπει όλοι να εφαρμόσουμε πολύ γρηγορότερα τις συστάσεις αυτές ε, να κάνουμε τις διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσεις πιο γρήγορα γιατί υπάρχουν εξωτερικά σοκ και το πώς αντιδράσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεγάλη σημασία για την απασχόληση στις 28 χώρες μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Χέι. Τον λόγο έχει ξανά ο εισηγητής. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους τους ε, συναλλεύσεις και οδησηγητές από άλλες πολιτικές ομάδες για τα σχόλιά τους, για τις παρατηρήσεις. Ευχαριστώ όλους που συμμετείχαν στη συζήτηση, γιατί όλα αυτά που ελέγχθησαν, κατά την άποψή μου, ε, είναι πολύ σημαντικά ε, θα βοηθήσουν την περαιτέρω συζήτηση επί της έκθεσης. Όπως είπαν λοιπόν ήδη μερικοί, Έχω την αίσθηση εδώ του αποκαλούμενου déjà vu, ότι μία από τα ίδια, γιατί ε, εμφανίζονται τα ίδια θέματα, τα ίδια λέμε, όπως και σε παλαιότερες συζητήσεις, ε, τότε που συζητάγαμε ε, για την έκθεση της ανάπτυξης σε αρχές του έτους. Εγώ βεβαίως δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες, κυρίως όσον αφορά τις επιπτώσεις της ε, λιτότητας ε, σε σχέση με την ύφεση, ούτε θα αναφερθώ στη σημασία των ε, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Καλύτερα αυτή τη συζήτηση να την αφήσουμε στις σχέσεις που θα έχουμε και συνεργασία για την προετοιμασία του τελικού σχεδίου. Όμως, επιτρέψτε μου να επισημάνω δύο-τρία πράγματα που ελέγχθησαν σε αυτή τη συζήτηση. Λοιπόν, Όσοι πιστεύουν ότι δεν αποδίδω αρκετή σημασία στα θέματα της ανεργίας ή της απασχόλησης, κοιτάξτε, νομίζω ότι το θέμα της ανεργίας αναφέρεται σε τουλάχιστον δύο-τρία σημεία της έκθεσης. Και μην ξεχνάτε ότι το αρχικό σχέδιο της έκθεσης ε, είναι περιορισμένο. Υπάρχουν εδώ κάποιες ρυθμίσεις. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να έχει στο σχέδιο πάνω από 4.000 ε, γράμματα, στοιχεία, Άρα δηλαδή είναι κανείς αναγκασμένος να κάνει περικοπές, να κάνει κάποιες ε, περιλήψεις, οι οποίες ε, περιλήψεις αυτές ε, δεν αντικατοπτρίζουν πάντα την άποψη του εισηγητή. Επίσης, να πω το εξής, αυτό το θέμα που έρχεται και επανέρχεται, το θέμα τις ε, σχέσεις ανάμεσα στις επενδύσεις και τις ε, περικοπές προϋπολογισμών. Νομίζω, έχω καταστήσει σαφές την έκθεσή μου ότι αν μια χώρα έχει αρκετό δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να στηρίζει τόσο τις δημόσιες όσο και ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτό το πλαίσιο, το περιθώριο το χρησιμοποιεί για να αναθερμαίνει την οικονομία. Αυτό είναι σαφές, αλλά δεν ισχύει αυτό για όλες τις ε, χώρες μέλη, γιατί <clears throat> ορισμένες εξαπτών εξακολουθούν να έχουν τεράστια προβλήματα λόγω δημόσιου χρέους. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να λαμβάνετε υπόψη. Τώρα, η περίπτωση της Ελλάδας είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Μπορούμε τώρα να ξεκινήσουμε πάλι μια μακρά συζήτηση, αλλά δεν νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Κατόπιν τούτου, ανακεφαλαιώνοντας, θα ήθελα για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω όλους όσοι παρενέβησαν και να επισημάνω ότι είμαι πρόθυμος ε, να συνεργαστώ με τους συναδέλφους μου και οδησίγητες για να βελτιώσουμε την έκθεση και για να καταλήξουμε σε ένα έγγραφο το οποίο θα αντικατοπτρίζει με το βέλτιστο δυνατό τρόπο πολιτικές και άλλες ε, ουσιαστικές ε, θέσεις όλων των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόεδρος, και εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Ρωσάτη και τώρα νομίζω ότι πρέπει να περάσουμε στο επόμενο θέμα της Μεσοδιάταξης, αλλά πριν περάσουμε σε αυτό θα ήθελα να σας υπενθυμίσω το χρονοδιάγραμμα για αυτήν την έκθεση 9 Σεπτεμβρίου, καταληκτική ημερομηνία για κατάθεση τροπολογιών. Οι τροπολογίες θα συζητηθούν στις 13 Οκτωβρίου και η ψηφοφορία στην Επιτροπή θα γίνει την ίδια μέρα. Και τέλος, η ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα γίνει ε, στη δεύτερη Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης στην ψηφοφορία. Ε, όμως ο κ. Γκολτιέρη θα προεδρέψει τις ε, ψηφοφορίες. Να περιμένουμε λοιπόν λιγάκι. Να δούμε τι θα κάνει ο κ. Γκολτιέρη. Αν δεν έρθει θα προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Πριν τις ψηφοφορίες, την ψηφοφορία έχουμε ένα άλλο σημείο, λέει ο πρόεδρος. Ah, έχουμε πράγματι να εξετάσουμε τις τροπολογίες της έκθεσης που θα ψηφίσουμε. Λάθος μου, με συγχωρείτε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Λοιπόν, εξέταση των τροπολογιών για το Γενικό Προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Οικονομικό Έτος 2016. Έχουμε τον εισηγητή κύριο Πέτερ Σίμων, παρακαλώ. Και συγγνώμη και πάλι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδης και όλους τους άλλους συναδέλφους της ΕΚΟΝ για τις ε, τροπολογίες, πολύ πολυάριθμες τροπολογίες που κατέθεσαν και για τη θαυμάσια συνεργασία που είχαμε για τη, στην αναζήτηση των ε, συμβιβασμών. Ε, όλα αυτά έγιναν το καλοκαίρι, δεν ήταν και αυτονόητο ότι θα πάνε τόσο καλά, γι' αυτό ευχαριστώ ιδιαίτερα. Τώρα, όσον αφορά του τους συμβασμούς στους καταλήξαμε, νομίζω ότι οι συμβασμοί αυτοί μας ε, οδηγούν σε μια πολύ πολύ καλή έκθεση. Καταλήξαμε σε συμβιβασμό, ο οποίος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία σε επενδύσεις και ανάπτυξη Συμβασμό Α. Τοποθετούμεθα επί το ΕΦΣΥ συμβασμός, Β και με συμβασμούς C, D και E και εκεί καταλήξαμε σε θαυμάσιους συμβασμούς όσον αφορά τη χρηματοδότηση των εποπτικών αρχών ε, του προσωπικού τους ε, και τι θα συμβεί και με το ρόλο αυτού του προσωπικού. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε τρία θέματα και αυτό το κάνω, ε, θα αναφερθώ μόνο σε αυτά γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Οι εποπτικές αρχές που αναφέρονται στις, ε, στο συμβασμό ήταν πολύ σημαντικές για μας και για τους σοσιαλδημοκράτες και χαίρομαι που καταλήξαμε σε ευρεία συνένεση γιατί πρέπει να σας πω για μένα εγώ φοβήθηκα, τρομοκρατήθηκα είχα προσωπικές συζητήσεις με αυτές τις εποπτικές αρχές και διαπίστωσα ότι παρότι υπάρχουν σημαντικές αυξήσεις στον προϋπολογισμό παρόλα αυτά έχουμε την ΕΜΠΑ, τη ΕΖΑ, την ΟΠΑ. Δεν θέλω τώρα να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά εν πάση περιπτώσει είχαμε ε, προσωπικότητες αυτών των αρχών οι οποίες ε, παρά τις αυξήσεις ε, δήλωσαν ότι δεν θα μπορούσαν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Δηλαδή τι έγινε, εμείς τους αναθέσαμε καθήκοντα, αλλά δεν υπήρχαν τα χρήματα για να κάνουν τη δουλειά τους. Ε, ο προπολογισμό του 16 θα πρέπει πρώτα απ' όλα να αλλάξει αυτό. Ένα άλλο σημαντικό θέμα για μένα είναι ε, αυτό που έχει σχέση με τις ε, προτεραιότητες στον τομέα του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εδώ λοιπόν είμαστε υπέρ της αύξησης του 4% στον προπολογισμό προσωπικού στον τομέα του ανταγωνισμού. Όποιος ανήκει στην Επιτροπή Τάξε γνωρίζει πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι αυτό. Γιατί ακούμε από κάποιους ε, ότι η περίπτωση McDonald's σε 16 εκατομμύρια ε, φόρους με ε, ένα απίθανο ποσό εισπράξεων το πώς εντοπίστηκε λοιπόν αυτή η περίπτωση η Κομισιόν δεν θα μπορούσε ποτέ να το εντοπίσει αυτό αν δεν υπήρχε αυτή η μελέτη των συνδικάτων. Όποιο λοιπόν το ξέρει αυτό, ε, τότε είναι αναγκασμένο και να διαρωτηθεί κατά πόσον η Κομισιόν με το προσωπικό που έχει αυτή τη στιγμή μπορεί να εκπληρώνει το ρόλο τη που είναι θεματοφύλακα των συνθήκων. Άρα δηλαδή οφείλουμε να στηρίξουμε ανεπιφύλακτα την Επιτροπή έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί με τους πόρους που διαθέτει. Και ειδικά στο θέμα της φορολογία να μεριμνήσει έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη αυστηρότητα ε, πρακτικές ε, καταστρατήγησης φορολογικών ρυθμίσεων. Περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Τελευταίο θέμα. Στην πρόταση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσβλέπεται αύξηση των οικονομικών πόρων στο Fiscalis 2020, βελτίωση της συνεργασίας των εθνικών φορολογικών αρχών. Το Συμβούλιο μείωσε την πρόσθεση κομισιών κατά 5 εκατομμύρια και χαίρομαι πάρα πολύ που καταλήξαμε σε μια συμβαστική πρόταση η οποία προβλέπει τον προσανατολισμό στην αρχική πρόταση της Επιτροπής, διότι η κακή ή ανύπαρκτη συνεργασία ανάμεσα σε φορολογικές, εθνικές φορολογικές αρχές είναι ένα από τα αίτια για το ότι στην Ευρώπη σε περίπτωση πολυεθνικών επανειλημμένα αναγκαζόμαστε να ομολογήσουμε ότι η φόρο αποφυγή είναι το αποτέλεσμα της έλλειψης συνεργασίας. Άρα δηλαδή πρέπει να χρηματοδοτηθεί επαρκώς το πρόγραμμα Φισκάλης 2020. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια ρύθμιση που θα βοηθήσει στη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Σκιώδης εισηγητές. Πρώτος ε, από το έλκο κύριο Ρωσάτη. Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Σίμων για την προετοιμασία της γνωμοδότησης και γιατί ήταν πάρα πολύ συνεργάσιμος σε ό,τι αφορά την κοινή μας δουλειά από των συμβαστικών προτάσεων. Εκτιμώ ιδιαίτερα αυτό το πνεύμα συνεργασίας και νομίζω ότι καταλήξαμε σε εύλογους συμβιβασμούς για τα περισσότερα επίμαχα σημεία. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να, υποστηρίξουμε τους συμβιβασμούς και ελπίζω και η ομάδα μου να ψηφίσει υπέρ της έκθεσης αυτής. Ίσως υπάρξουν ε, ε, αρνητικές ψήφοι για κάποιες μεμονωμένες τροπολογίες, αλλά αυτές δεν προέρχονται τη δική σας πολιτική ομάδα. Να σας συγχαρώ για μια ακόμη φορά και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε με την έκθεση αυτή. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ρωσάτη εκ μέρους ε, της ομάδας ECR, η κυρία Κέ Σουίμπορν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για το ότι λείπει η σκιώδη συγγήτρια του ECR για να ευχαριστήσει τον εισηγητή για τη σκληρή δουλειά που έκανε. Θα ήθελα να εξηγήσω λοιπόν πως η θέση μας πάνω σε αυτό το θέμα δεν οφείλεται στη σκληρή δουλειά του εισηγητή που έκανε βέβαια σκληρή δουλειά αλλά στην πάγια θέση μας υπέρ τη δημοσιονομικής πειθαρχία. Εμείς δεν θεωρούμε πως όλο ένα αυξανόμενο προπολογισμό θα βοηθήσει την Ένωση και οποιαδήποτε αύξηση σε δαπάνε πρέπει να αντισταθμίζεται με μείωση σε άλλον τομέα. Αυτή είναι η θέση μας ε, στο σύνολο του προπολογισμού. Γι' αυτό τον λόγο δυστυχώ δεν μπορούμε να στηρίξουμε τι ε, περισσότερε τροπολογίε τη ΕΚΟΝ. Δεν υπάρχει ε, λογική για να μπορέσουμε να σκεφτούμε εναλλακτικές στην αύξηση της χρηματοδότησης. Και βεβαίως αντιλαμβανόμαστε την πάρα πολύ μεγάλη δουλειά που γίνεται και όταν υπάρχουν τόσο μεγάλοι περιορισμοί στους προϋπολογισμούς σε όλη την Ένωση δεν μπορούμε να δεχτούμε ε, περαιτέρω αυξής του προπολογισμού και θα πρέπει να βοηθεί το έργο του προπολογισμού της ε, ΙΣΑ. Σας ευχαριστώ ο κύριος για τους ε, φιλελεύθερους. Δεν είναι εδώ. Δεν ξέρω αν κάποιος από το Άλντε θα... κάτι. Γκουε. Α, ο κύριος Μπέγκας. Αν με επιτρέπετε, θα ήθελα να κάνω κάποιε παρατηρήσει για τον προπολογισμό αυτό που ουσιαστικά εκφράζει ε, τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όπως ε, υπόθηκε και εδώ, δείχνει ε, μία διαφορά μεταξύ των προθέσεων και των μέσων που διατίθεται για την υλοποίηση αυτών των προθέσεων. Με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να επιτευχθούν αποτελεσματικά οι πολιτικοί στόχοι που έχουν ανακοινωθεί. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Για, τα, για την επιτήρηση ε, και την εποπτεία. Νομίζω ότι υπερβάλλουμε ως προς τα αποτελέσματα τα θετικά μπορεί να έχει. Δεν βλέπουμε σε αυτό τον προϋπολογισμό και είναι μια γενική παρατήρηση αυτή. Δεν βλέπουμε λοιπόν τα απαραίτητα μέσα για να αντιμετωπιστεί το εύρος της κρίσης στην οποία, την οποία βιώνουμε. Δεν βλέπουμε να έχουν υιοθετηθεί τα απαραίτητα μέτρα για να λυθούν τα προβλήματα που προκαλεί η κρίση. Όπως είναι οι ασυμμετρίες που υπάρχουν ε, εντό της Ένωσης. Πολύ καλό είναι το επενδυτικό πρόγραμμα, γιατί όχι ε, μιλώντας, γιατί το συγκεκριμένο επί του περιεχομένου ε, δεν μπορώ να πω ότι με βρίσκει απόλυτα σύμφωνα, αλλά ο προπολογισμό. Δεν θα πρέπει να στρέφεται σε άλλα θέματα πλην λιτότητα και απορρίθμιση. Δεν θα πρέπει να προσπαθεί να βρει λύσει στην κρίση του δημοσίου χρέους. θεωρούμε ότι χρειάζονται πολύ περισσότεροι πόροι για να αντιμετωπιστούν τα πραγματικά προβλήματα που δεν έχουν να κάνουν τόσο με την εποπτεία όσο με την καταπολέμηση της ε, κρίσης. Και στο συγγνώμη αν ε, σας φαίνομαι απεσιόδοξος, αλλά βλέπω μια τεράστια ε, διαφορά μεταξύ προθέσεων και πραγματικών μέσων. Ευχαριστούμε λέει ο Πρόεδρος τώρα από τους πρασίνους ο κύριος Γκίγκολτ. Thank you, Pablo. Ευχαριστώ, Παύλο. Πρώτα απ' όλα, ε, ευχαριστώ τον εισηγητή. Πρόκειται για μια πάρα πολύ καλή έκθεση. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια, ούτε γενικές ομιλίες για το πώς πρέπει να σχεδιαστεί ο προϋπολογισμός της Ένωσης ε, δεν μπορούμε εδώ να εξοικονομήσουμε ε, πολλά λεφτά ούτε τώρα είναι η στιγμή να μιλήσουμε για τεράστια αύξηση του προϋπολογισμού όλα αυτά είναι σημαντικά αλλά δεν είναι ε, τώρα η στιγμή που πρέπει να συζητηθούν είναι καλή έκθεση στέλνουμε τα σωστά μηνύματα και δίνουμε τα χρήματα που χρειάζονται στο Ευρωπαϊκό Εποπτικό Σύστημα και το να λέμε απλά το ότι χρειαζόμαστε περισσότερο προσωπικό από τα κράτη-μέλη δεν θα λύσει τα προβλήματα. Ποιος έχει πάει στα θεσμικά αυτά όργανα ξέρει ποια είναι τα προβλήματα και πρέπει να τα πάρουμε σοβαρά αντί να κάνουμε γενικές ε, παρατηρήσεις ε, για την ε, δημοσιονομική πειθαρχία. Όταν μιλάμε λοιπόν για τις δαπάνες, καλό είναι να δώσουμε δύο μηνύματα. Το ένα είναι πως ε, το, εάν η ΆΙΖΑ πάρει τα λεφτά μας θα πρέπει να φροντίσουν η πρόσβαση στα έγγραφα για τα κοινοβούλια να είναι εξίσου καλή με αυτή που δίνουν στους λομπίστες και τα κράτη-μέλη και πρέπει να δούμε ξανά τις δημοκρατικές αρχές στα συστήματα ΕΦΡΑΚ και ISB όπου εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη δημοκρατικών αρχών, κάτι το οποίο βεβαίω δεν συνάδει με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ευχαριστώ λοιπόν πάλι τον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές για την καλή συνεργασία. Ευχαριστώ. Από το EFD δεν υπάρχει κανεί Και δεν ε, έχω εδώ κάποια επιβεβαίωση. Δεν ξέρω αν Θέλει κάποιο λόγο από τη νέα ομάδα. Περνάμε λοιπόν στο KTI. Ο κ. Μαριάς έχει ζητήσει το λόγο. Πρόεδρε, θα πάρω αφορμή από την τροπολογία 6319 που αφορά τις δαπάνε για το μηχανισμό συμβολή στη σταθερότητα και την ειρήνη. θέλω να πω ότι ο προϋπολογισμός μας πρέπει να λάβει σοβαρά πλέον υπόψη τα τεράστια προβλήματα που δημιουργούνται για τις χώρες της Μεσογείου κυρίως, στην Ελλάδα, την Ιταλία αλλά και άλλες χώρες, από το τεράστιο κύμα των προσφύγων και των παράνομων μεταναστών που έρχονται πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να το ξεκαθαρίσουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί, ιδίως από τη Συρία και άλλες εμπόλεμες περιοχές, φεύγουν προκειμένου να γλιτώσουν τη ζωή τους. Και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει σαφέστατες παρεμβάσεις προκειμένου να εμπεδοθεί η ειρήνη ιδίως στις ε, χώρες της ε, Μέσης Ανατολής και στην Αφρική όπου υπάρχουν ε, τεράστιες συγκρούσεις. Διαφορετικά θα έχουμε συνεχώς τεράστια κύματα προσφύγων. Άρα λοιπόν είναι σημαντική η παρέμβαση η ειρηνευτική στις περιοχές αυτές. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να βοηθήσει και την ανάπτυξη των περιοχών αυτών για να έχουμε λιγότερους ε, παράνομους μετανάστες. Όλα αυτά χρειάζονται κονδύλια και μια τελείως διαφορετική ε, διάρθρωση του προϋπολογισμού. Τέλος, να σας ενημερώσω, αλλά θα το έχετε δει, ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση με τις ε, προσφυγικές ροές στην Ελλάδα έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της. Σας λέω ότι ο δήμαρχος της Λέσβου, της Μητυλίνης έστειλε μια επιστολή να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έχει 85.000 κατοίκους η Λέσβος σήμερα και υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλούμε πάνω από 10.000 πρόσφυγες και παράνομοι μετανάστες μέσα στην πόλη της Λέσβου. Είναι αδύνατο να γίνει πλέον από την πλευρά της Ελλάδας διαχείριση αυτών των μεταναστευτικών και κυρίως προσφυγικών ροών. Το καλοκαίρι ήμουνα στη Σάμο. Όλο το νησί ήταν γεμάτο από πρόσφυγες οι οποίοι είχαν έρθει από την Τουρκία και πήγα στην Τουρκία να δω τι γίνεται. Δεν βρήκα ούτε ένα πρόσφυγα ή μετανάστη να κυκλοφορεί στο Κουσάνταση. Πού βρίσκονται όλοι αυτοί και ξαφνικά την επόμενη μέρα επιβιβάζονται οργανωμένα σε λέμβους μεσοσύβια και φτάνουν στα νησιά του Αιγαίου. Είναι δεδομένο ότι πρέπει να γίνει παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Τουρκία, διότι από εκεί γίνεται ένα δουλεμπόριο και έρχονται όλοι οι πρόσφυγες οι οποίοι πραγματικά είναι σε απελπιστική κατάσταση. Αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί παρά μόνο πολιτικά. Αλλά επίσης τα κονδύλια που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα είναι ψίχουλα. 70 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Δεν αρκούν. Άρα λοιπόν σας το επισημαίνω αυτό ότι πρέπει η λογική του προϋπολογισμού να λάβει σοβαρά υπόψη αυτή τη νέα πίεση που υπάρχει στην Ελλάδα, στην Ιταλία και σε ορισμένες άλλες χώρες. Διότι μόνο όταν υπάρξει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και κονδύλια σοβαρά μπορούν οι χώρες αυτές να υποδεχτούν, αν μπορούν να υποδεχτούν, αυτό το τεράστιο κύμα των προσφύγων. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι γεμάτη ανέργους, φτώχεια. Δεν μπορεί να έχει πλέον άλλους πρόσφυγες και παράνομους μετανάστες. Να το καταλάβετε αυτό. Άρα λοιπόν λέω κύριε Πρόεδρε ότι πρέπει με αφορμή αυτή την τροπολογία την 6319 που προβλέπει κονδύλια να υπάρξει μια άλλη φιλοσοφία στον προϋπολογισμό αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε σοβαρά αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται μια άλλη αντιμετώπιση στα ζητήματα αυτά. Ευχαριστώ. Thank you very much uh, Mr. Marias. Now I give the floor to Mr. Thomas Mann. Σας ευχαριστώ, ο κύριος Thomas Mann. Um, Ευχαριστώ πολύ. Ε, κοιτάξτε, αυτή η τελευταία παρατήρηση ήταν απόλυτα σαφής. Όταν συζητάμε για τον προεπλογισμό σε διάφορα κράτη-μέλη, αυτή είναι μια πολιτική συζήτηση ε, που γίνεται, αλλά κατ' ουσίαν πρόκειται για αυτό που είπε ο Πέτερ Σίμων ε, και το έκανε πολύ καλά, συγκεκριμένοι αριθμοί, Πού υπάρχουν προβλήματα. Εμεί ε, είμαστε Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. σαφώ και μπορούμε να ασχοληθούμε και του πρόσφυγες, αλλά υπάρχουν και άλλε επιτροπέ, α πούμε στην Επιτροπή απασχόληση. εκεί εστιάσαμε την προσοχή μα σε αυτό το θέμα. Δεν μπορούμε με βάση ένα θέμα, μία γραμμή του προπολογισμού να πούμε αμφισβητούμε όλο τον προπολογισμό. Και το θέμα των προσφύγων δεν είναι μόνο θέμα πόρων και χρημάτων, είναι και κατά πόσο είμαστε σε θέση ε, να ε, δημιουργήσουμε δομέ. Και συνάδελφε, την Τετάρτη θα τα πούμε ο κύριος Γιούγκερ θα έρθει για να μας πει τι θα γίνει με τους πρόσφυγες. Και κοιτάξτε, δεν θα υπάρχουν δηλώσεις προθέσεων, αλλά θα εξετάσουμε νομοθετήματα, συγκεκριμένα λοιπόν μέτρα για να επέλθουν αλλαγές και το θέμα της ε, παρατυπίας και παρανομίας ε, μεταναστών, θέμα διακινητών, συγκεκριμένα δηλαδή. Εκεί να τα κουβεντιάσουμε. Αλλά τώρα νομίζω ε, καλύτερα να δούμε λιγάκι του αριθμούς. Τώρα ε, παίζουν ρόλο οι αριθμοί και χαίρομαι που ο κύριος Ζήμων ε, ε, έχει μια πολύ καλή έκθεση συνεργασία με τους εισηγητές, βεβαίω και είναι διαφορετικέ οι προτεραιότητες και πρέπει να ελέγξουμε καλά τον προπολογισμό. Συνάδελφοι από την Ελλάδα, σε εσά απευθύνομαι, θα πρέπει να μεριμνήσουμε έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί να χρησιμοποιήσει το άρθρο 78 και αν μπορεί κανείς να κάνει κάτι θα διαθέσουμε τους απαραίτητους πόρους. Το άλλο, καλά το είπατε, είναι πολιτική φύση το θέμα και πρέπει να εξεταστεί αλλού. Άρα δηλαδή χαίρομαι ότι ε, έχουμε αυτή τη συζήτηση και ελπίζω να έχουμε και πλειοψηφία για την έκθεση που μας υποβλήθηκε. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Ε, δίδω τώρα και πάλι το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Πίτερ Σάιμον. Σας ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Εντάξει, είχε κάποιες διαφοροποίησεις. Ευχαριστώ που με πενέσατε κιόλας. Η συνεργασία ήταν πολύ καλή. Ε, σε άλλους, σε τους μήνες που πέρασαν, δεν κατέστηναν τι. Σε εμάς πήγε πολύ καλά. Αναφέρομαι τώρα στην κριτική του συναδέλφου ότι θα πρέπει να αναφερθούμε περισσότερο στην τροπολογία 63-19 και το αιτιολόγησε με την προβληματική των προσφύγων. Κοιτάξτε, η τροπολογία αυτή και κυρίως η αιτιολογία της, επουδενή δεν πρέπει να δώσει λαβή το να σκεφτεί κανείς ότι αυτό το θέμα έχει απαραίτητα σχέση με τις πρόσφυγες. Και σας διαβάζω την αιτιολογία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενισχύσει την ταυτότητά της ως ένα υπεριαλιστικό στρατιωτικό μπλοκ. Έχει εμβαθυνθεί η στρατιωτικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το καθεξής. Δηλαδή, στην αιτιολογία πρόκειται για κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που συζητάμε σήμερα. Και γι' αυτό, όπως είπε και ο συνάδελφος Μαν, εγώ περιορίστηκα στα θέματα που αφορούν την ΕΚΟΝ. Τώρα, τα στρατιωτικά και άλλα, αυτά δεν είναι δική μας δουλειά. Οι πρόσφυγες ε, το ότι κρύβονται αυτοί πίσω από αυτή την τροπολογία, ειλικρινά σα λέω αγαπητέ συνάδελφε, αυτό κανεί δεν το σκέφτηκε. Κανεί. Κανενό το μυαλό δεν πήγε στου πρόσφυγες. Λοιπόν, άλλη παρατήρηση στο case Wimburn. Βεβαίως και καταλαβαίνω ότι υπάρχουν δυσκολίε για αυξήσει ε, σε συγκεκριμένου τομεί, αλλά κυρίω σε όλους εκείνου του τομεί, όπου τα τελευταία χρόνια υπήρξε μεγαλύτερη εποπτεία έτσι ώστε στο μέλλον αν θέλετε να αποφύγουμε μια παρεμφερή χρηματοδοτική κρίση ή να δημιουργήσουμε εμπόδια για να προκύψει τέτοια κρίση, τα εμπόδια αυτά να είναι πιο ουσιαστικά. Αυτά τα εμπόδια λοιπόν για αναχέτηση κρίσης υπάρχουν, αλλά τι λείπει, λείπει το προσωπικό και γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι καθήκον αυτού του Κοινοβουλίου και της ε, τρέχουσας θητείας να σταθεροποιηθούν αυτά, αυτή η αναχαιτιστική φραγμή τα φράγματα που θα αντιμετωπίσουν τη θύελα. Και ε, όταν οι αρμόδιες εποπτικές αρχές λένε δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας, δεν έχουμε προσωπικό, αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Γιατί αν δεν το κάνουμε θα είμαστε συνένοχοι αν την επόμενη φορά που ενδεχομένω να προκύψει κρίση, ναι εντάξει καλά θα τα έχουμε ρυθμίσει στα χαρτιά για τις εποπτικές αρχές, στην πράξη όμως δεν θα έχουμε πετύχει τίποτα. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σάιμον. Έτσι λοιπόν τώρα θα ψηφίσουμε, λέει ο πρόεδρος. Κύριε Μαριά. Ε, one minute, please. seconds. One, okay. <laughs> Every time. Ε, ήθελα να επισημάνω το εξή. Εγώ αναφέρθηκα στην τροπολογία δαπάνε στήριξη για το μηχανισμό συμβολή στη σταθερότητα και την ειρήνη για να επισημάνω ότι χρειάζονται οι δαπάνε στήριξη. Δεν υποστήριξα και δεν είπα ότι ψηφίζω υπέρ της τροπολογίας που αφαιρεί τα ποσά αυτά με ένα σκεπτικό. Εγώ λέω ότι πρέπει να παραμείνει η γραμμή αυτή, διότι η τροπολογία λέει να φύγει. Εγώ λέω να παραμείνει η γραμμή αυτή και να αντιληφθούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ενίσχυση δαπανών για την συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ειρήνη, ιδίως σε περιοχές που ανέφερα της Μέσης Ανατολής, για να μην έχουμε κύματα προσφύγων προς την Ελλάδα, προς την Ιταλία. Σας επισημαίνω ότι 130.000 νέοι πρόσφυγες ήρθαν στην Ελλάδα από τις αρχές του έτους. Πολύ περισσότεροι από ό,τι έχουν πάει στην Ιταλία. Άρα είπα το ακριβώς αντίθετο κύριε Σιγητά. Ευχαριστώ. Thank you. Mr. Simon, you have the floor. letzter Kommentar dazu ein τελευταία μου παρατήρηση, κοιτάξτε, μια τροπολογία η οποία ε, προβλέπει αύξηση δεν έχει κατατεθεί, δεν έχει κατατεθεί η τροπολογία, τώρα, άρα δεν μπορούμε να ψηφίσουμε από αυτή σήμερα. Πρόεδρος, πάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ψηφοφορία, αλλά όπως είπα και προηγουμένως, ο κύριος Γκουαλτιέρη θα ε, προεδρέψει, μόλις έρχεται ο κύριος ε, Γκουαλτιέρη, θα του, παραδώσω την έντρα. Ευχαριστώ. Dear colleagues, good morning. I hope uh, Καλημέρα αγαπητοί Good holidays. Ελπίζω να περάσετε καλά, καλές διακοπές. Ε, ξανά στη δουλειά τώρα. Έχουμε την πρώτη μας ψηφοφορία. Το σχέδιο γνωμοδότης για το Γενικό Προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισηγητής μας ο κύριος ε, Πέτερ Σίμων. Και ξεκινάμε με ένα έλεγχο Παρακαλώ τους συναδέλφους να τοποθετήσουν ε, στο μηχάνημα της κάρτας ψηφοφορίας και τώρα ξεκινά η δοκιμαστική ψηφοφορία. Ah, Still three colleagues to vote. Τρεις συνάδελφοι δεν έχουν ακόμη ψηφίσει. Okay, we close the vote. Ωραία, η ψηφοφορία. Αν κάποιος δεν έχει μαζί του την κάρτα να μας το πει, όλοι έχετε τις κάρτες σας πάρα πολύ ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν με τις δημοσιονομικές τροπολογίες. Όχι με το ψήφισμα. απολογια ΕΚΟΝ 6315. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6314. Χωριστή ψηφοφορία. Μάλλον σε τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι γκρίνεται. Ας ελέγξουμε όμως καλύτερα. Άρχεται η ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα. Από τους σοσιαλδημοκράτες ένας παραπάνω. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. ΠΕΡ, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Έκον 63-16. Όχι. Ναι. 63-16. Ψήφι ΠΕΡ, Κατά αποχες 634 υπέρ κατά να ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία πέρασε απορρίπτεται 63-23. Ψήφι περ. Κατά αποχές εγκρίνεται 63-13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 63-02 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 63-17 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 63-11 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε την 63-11. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Απορρίπτεται με ισοψηφία. 63-05 λοιπόν. Πάντα σε τροπολογίε από το προπολογισμού. Υπέρ, κατά, αποχέ. Εγκρίνεται. 63-05. 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 6309 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 6303 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 6307 υπέρ κατά νομίζω απορρίπτεται να ελέγξουμε την 6307. Disclose. τη της Απορρίπτεται. 63-10. Άρχεται, μάλλον ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 63-12. Υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε την 63-12. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 63-25. Υπέρ κατά απορρίπτεται αλλά μήπως να ελέγξουμε καλύτερα άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται πράγματι 6306 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6318 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6319 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 6322 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 6300 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 6321 υπέρ, Όχι, πάμε στην 6320 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 6308 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ευχαριστώ. Τελειώσαμε τις τροπολεύσεις του προπολογισμού και πηγαίνουμε τώρα στην γνωμοδότηση, στο σχέδιο γνωμοδότησης. Συμβιβαστική α υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά να την επαληθεύσουμε λοιπόν την 5, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Απολογία 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ, κατά νομίζω πως απορρίπτεται. Να την επαληθεύσουμε την 7. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική Β υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 18 υπέρ. 20 με συγχωρείτε υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 21 υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία πέρας να απορρίπτεται 22 υπέρ κατά να απορρίπτεται 23 υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική γάμα υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Η 29 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 31 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε την 31 άρχεται τη ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται συμβαστική δέλτα υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 35 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε πάλι 35 πέρας Αχα, απορρίπτεται. Μάλλον χρειάζομαι γελιά καινούρια. Συμβαστική α υπέρ, ε, ε, ε, ε υπέρ κατά έχει ε, δεκτεί. Τροπολογία 39 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 υπέρ κατά, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 42 υπέρ κατά αποχές δεκτή 43 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική F υπέρ κατά αποχές δεκτή G υπέρ κατά αποχές δεκτή αρχικό κείμενο παραγραφός 10 υπέρ όχι έχει αποσυρθεί ναι αλλά το αρχικό κείμενο άρα παραμένει άρα το ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο της παραγράφου 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή Τροπολογία 52 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 53 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 54 υπέρ. Κατά. Νομίζω πως απορρίπτεται. Να την επαληθεύσουμε όμως άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή με μία ψηφοδιαφορά. 55 υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία πέρασε δεκτή και τώρα ψηφίζουμε το κείμενο όπως τροποποιήθηκε υπέρ με ηλεκτρονική ψηφοφορία με συγχωρείτε άρχεται η ψηφοφορία 40 υπέρ, 12 κατά, μία εποχή εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Επόμενη συνεδρίαση, Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, με τον κύριο Δράγκη κιόλας. Καλά τα λέω. Τρίτη. Τρίτη, και 3η 15 Σεπτεμβρίου πρωί και απόγευμα θα σας στείλουμε την ημερήσια διάταξη. Ελίζα, θέλεις να πεις κάτι. Να ζητήσω η γραμματεία ή δυνατόν ε? να βάλει το αρχικό του ονόματός μου μπροστά στο επιθετό μου. Δεν ήμουν εγώ η Φερέιρα, αλλά ο Αλφαζάν Ζαν Φρέιντα γιατί είναι δύσκολο αν δεν υπάρχει και το αρχικό γράμμα του ονόματος μπερδευόμαστε έχουμε το ίδιο επίθετο ναι γιατί και εγώ σας έβλεπα να ψηφίσετε κατά του ίσως του αυτού λέει ο πρόεδρος και είχα ε, εκπλαγεί τώρα κατάλαβα μάλιστα ωραία έχετε δίκιο πρέπει να, να το διευκρινίσουμε πέρα συνεδρίσεις